Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στηρίζω αυτό το ψήφισμα που προτείνουν πολλές πολιτικές ομάδες και πιστεύω και εγώ ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των πολιτών μετά τη Συμφωνία Αποχώρησης δεν πρέπει να σπάσουν οι παλιοί δεσμοί. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα τα δικαιώματα αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα των Βρετανών αλλά και των υπόλοιπων Ευρωπαίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε πολλά επίπεδα. Το κράτος δικαίου αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπώς οφείλει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα περισσότερο από ποτέ. Είναι ένα ηχηρό μήνυμα που πρέπει να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες των πολιτών και ότι δεν φτάνει ένα αυτόματο σύστημα καταχώρησης. Τα δικαιώματά τους παρακαλώ να τα προστατεύσετε. Ευχαριστούμε. Χουκ τώρα εκ του Renew. Τόσα εκατομμύρια άνθρωποι από τις 27 χώρες ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι, νοσοκόμοι, γιατροί, άνθρωποι που φροντίζουν, εργαζόμενοι γενικά. Είναι φίλοι μας, είναι γειτονέ μας. Ε, κάποιοι από αυτού είναι και σύζυγοί μας. Οπότε πραγματικά μένω με το στόμα ανοιχτό με αυτές τις γραφειοκρατίες που εφαρμόζονται. Ε, είναι κάτι που προσβάλλει το αίσθημα δικαιοσύνη των ίδιων των Βρετανών. Τι κυβέρνηση κάνει του ανθρώπου οι οποίοι για χρόνια ζούσαν στη χώρα, που έχουν συνεισφέρει στην κοινωνία, με νόμου που του επέτρεπαν να πρέπει τώρα να ζητάνε την άδεια για να παραμείνουν και να του ζητάνε έγγραφα τα οποία δεν έχουν στη διάθεσή του. Υπάρχουν 90% των θέσεων ε, που υποβάλλονται και που πολλές από αυτές ε, περνάνε. Πρέπει λοιπόν μετά από τέσσερα χρόνια που έχουμε μείνει στα ίδια επίπεδα χωρίς να κουνιέται τίποτα, δεν πρέπει τώρα να πάμε στην καταστροφή. Ευχαριστούμε. Μπάιντεκ εκ μέρου της Ρινιού επίσης. Παρακαλώ. Είναι λυπηρό που σήμερα στο Κοινοβούλιο πρέπει να περάσει ένα ψήφισμα για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολυάριθμων Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών που ζουν στο εξωτερικό. Παρότι καλωσορίζω το ότι εγκρίναμε αυτό το ψήφισμα, τέτοια δικαιώματα δεν έπρεπε να διακυβευτούν ποτέ από τη Βρετανική κυβέρνηση λόγω του Brexit. Το πρώτο που έπρεπε να είχε κάνει η Τερέζα Μέη ήταν να εγγυηθεί τα δικαιώματα των Ευρωπαίων που ζουν στη Βρετανία. Θα τη έδινε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση και θα είχε απαλλάξει πολύ κόσμο από χρόνια στρε και αβεβαιότητα. Τώρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο εξαρτάται από ένα PDF ως απόδειξη ε, κατάστασης παρά οποιοδήποτε κάρτα ή χαρτί. Ένα PDF, όπως ξέρουμε, μπορεί να παραποιηθεί εύκολα, οπότε οι εργοδότες, οι ε, ιδιοκτήτες κατοικιών φυσικά ανησυχούν ε, για παραποίηση εγγράφων και αυτό θα οδηγήσει σε διακριτική μεταχείριση. Ελπίζω η Βρετανική κυβέρνηση να παραποιηθει ευκολα οποτε οι εργοδοτες οι ιδιοκτητες κατοικιων φυσικα ανησυχουν για παραποιηση εγγραφων και αυτο θα οδηγησει διακριτικη μεταχειριση ελπιζω η βρετανικη κυβερνηση να εισακουσει τις ανησυχίες των ανθρώπων ε, και να λάβει υπόψη το ψήφισμα το σημερινό. Αλλά και οι Βρετανοί πολίτε ανησυχούν σωστά για το δικαίωμά τους να παραμείνουν σε ευρωπαϊκέ χώρες που είναι σήμερα το σπίτι του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη που πρόσφεραν γενναιόδορε ε, προϋποθέσεις εγκατάσταση, ήδη στους Βρετανού πολίτε εκείνους που είναι μόνιμοι κάτοικοι στι χώρε αυτέ και παροτρύνω τι χώρε που δεν έχουν ακόμα δηλώσει τι προθέσει του να το πράξουν ε, και να ανακοινώσουν τι προθέσει του εν ευθέτω χρόνο. Επόμενη, ε, ομιλητή, ο Τζον Χάουαρθ. Όχι, κυρία Μπρόφη, όπω είπε η πρόεδρο, ανακοινώστε το λάθο άτομο. Είμαι ο Τζον Χάουαρθ. Το ψήφισμα αναφέρεται στη συμφωνία αποχώρηση ω ισορροπημένο έγγραφο, παρότι δεν είναι. Αν ήταν, δεν θα χρειαζόταν να περάσουμε τις τροπολογίες. Στην πραγματικότητα, οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δίκιο να φοβούνται, διότι το βρετανικό σύστημα, όπω λειτουργεί το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι συνταγματικά ρατσιστικό και θεσμικά ξενοφοβικό. Οποιοδήποτε ποτέ ασχολήθηκε με τέτοιες υποθέσεις το γνωρίζει. Επίσης είναι λάθος ε, ο τερματισμός τη ελεύθερη κυκλοφορία Είναι μια αρπαγή ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους πολίτες και οι Βρετανοί πολίτες που έχουν μεταναστεύσει στην ε, ε, υπηρετική Ευρώπη για να φτιάξουν μια ζωή εκεί βλέπουν ε, αποφάσεις ζωής να υπόκεινται σε ένα καθεστώς το οποίο αλλάζει η απόφαση μιας ψηφίας του Βρετανικού πληθυσμού. Είναι ντροπή. Στο ψήφισμα αυτό πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα πριν ψηφιστεί η συμφωνία αποχώρηση. Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε δεν πρόκειται μάλλον να υποστήριξω τη συμφωνία αυτή. Η κυρία Τζιν Πρόφη τώρα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα αυτό το κείμενο ε, Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ε, τρία ε, σημεία για πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων στην Αγγλία και Άγγλων στην Ευρώπη γιατί πάρα πολλοί δεν είχαν κάνει μέχρι τις 36 του 21 την αίτηση. Όποιος δεν την κάνει μέχρι τότε πρόκειται να εκδιωχθεί από τη χώρα και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ε, λέει το κείμενο ότι θα πρέπει όποιο είναι να έχει ένα χαρτί που να αποδεικνύει νόμιμη διαμονή και όποιος δεν το έχει τότε οι Ευρωπαίοι που είναι στην Αγγλία ε, θα κινδυνεύουν με μέτρα δεσμένους διάκρισης και έχουμε την απόφαση του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ε, αποχώρηση και χρειάζεται βέβαια για να κλείσει αυτή η συμφωνία να διασφαλίσει σχετικά με τα δικαιώματα αυτών των προσώπων το Ινωμένο Βασίλειο. Οπότε χρειάζονται κάποια μέτρα για την ασφάλεια δικαίου που θα αφορούν και τους Βρετανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ο επόμενος. Η Μπάρμπαρα Γκίμψον και εκείνη από τους Ρενιού. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι 100% πεπισμένη. Η απόφαση αποχώρησης είναι ένα τεράστιο σφάλμα. Πάντως, εάν υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τα δικαιώματα των Ευρωπαίων στην Αγγλία να προστατευτούν. Εκείνοι που μένουν στον Βασίλειο, αλλά επίση και οι κάτοικοι του Βασιλείου στις άλλες χώρες, οπότε σήμερα είδαμε πόσοι στο Κοινοβούλιο ενέκραναν αυτό το κείμενο που απετέλεσε μήνυμα προς την Βρετανική κυβέρνηση. Η προσέγγιση τους είναι ανεπαρκής γιατί τίποτα δεν θα κερδίσουν αν χρησιμοποιούν τον κόσμο σαν ατούστη στη διαπραγμάτευση. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο το ότι αποχωρούμε από την Ένωση, αλλά με χαρά μου ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου που κατοχυρώνει τα δικαιώματα του κόσμου σε σχέση με την αποχώρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Στάνισλαφ Πόλτσακ τώρα, εκ μέρου του ΕΛΚ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, εσείς κυρία Φόξ πρώτα. Ευχαριστώ, εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα. Γιατί πάντα το έλεγα από τότε που έγινε το 16 το δημοψήφισμα ότι οι πολίτες που θέλουν να μείνουν στο Ενωμένο Βασίλειο πρέπει να έχουν δικαιώματα πρέπει να τους προσφερθεί καθεστώς μόνιμης κατοικίας. Τώρα όμως εδώ επικρίνεται η κυβέρνηση για τους λάθος λόγους και ανοίγει μια διαδικασία που δεν θα έπρεπε να κάνει ε, βάσει δήλωσης. Δεν πρόκειται για καμιά απόδειξη και είναι γελίο αυτό. Έτσι, η κυρίαρχες κυβερνήσεις δεν μπορούν να ελέγξουν τι κάνουν μέσα στα σύνορά τους. Επίσης πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό έχει πολιτικοποιηθεί υπερβολικά γιατί συμπεριλαμβάνει και την ιδέα ότι η ελεύθερη διακίνηση είναι μια μεγάλη απώλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, αλλά βλέπετε έτσι μπαίνετε στο μάτι αυτών οι οποίοι ψήφισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς γιατί δεν θέλουν την ελεύθερη αυτή διακίνηση δεν πρόκειται για ξενοφοβία, δεν πρόκειται για εχθρική στάση απέναντι σε Ευρωπαίους πολίτες που έρχονται να επισκεφθούν, να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, λάθος. Πρόκειται για τον έλεγχο των συνόρων. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο της κυριαρχίας. Και εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτούς που έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις και όσοι θέλουν από τις ευρωπαϊκές χώρες να γίνουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευπρόσδεκτοι να το ζητήσουν και να γίνουν. Ευχαριστούμε. Τώρα Στάνισλαβ Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, ε, λυπούμε που βλέπω να αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την κοινότητά μας. Θα μπορούσαμε ίσω να ήμασταν πιο ισχυροί. Κάποιες χώρες μπορεί να χαίρονται, ξέρω εγώ, η Ρωσία, οι άλλε υπερδυνάμει. Πάντω εγώ καλωσορίζω την συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχει αυτή η συμφωνία, η οποία είναι ισορροπημένη, πιστεύω και στη μεταβατική περίοδο διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη, τη μελλοντική περίοδο, η συμφωνία μιλάει για υποχρέωση για μια σταθερή και ισορροπημένη και δίκαια λύση. Πρόκειται βέβαια για μια δήλωση. Πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και που δεν καλύπτονται ακόμα από τη συμφωνία. Μην ξεχνάμε τους ε, Σκοτσέζους ε, και άλλους. Είναι καλό πάντως που υπάρχει μια συμφωνία, γι' αυτό και τη στήριξε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μαρτίνα Άντερσον τώρα. Πριν από τις 31 Ιανουαρίου, όταν θα με πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τι δημοκρατικά πεπεφρασμένε άποψει των ανθρώπων του Βορρά που ψήφισαν υπέρ τη παραμονή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ευρωβουλευτέ που μαχήθηκαν και υπερψήφισαν το ψήφισμα σήμερα και για την υποστήριξή σα για τη Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή και όλα του τα κομμάτια. Αυτό το ψήφισμα ασχολείται με τα δικαιώματα των Ιρλανδών πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία για να απολαύουν την πρόσβαση και να μπορούν να ασκήσουν τα ευρωπαϊκά δικαιώματα όπου αποφασίσουν. Η Βρετανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε να αλλάξει τους ε, κανόνες μετανάστευσης. Όσοι έχουν γεννηθεί στη Βόρεια Ιρλανδία δεν θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους επανένωση οικογενειακή. Η Βρετανία όμως ε, ονομάζεται ε, ε, για κάποιους λόγους. Όσοι έχουμε γεννηθεί στη βορεια θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε Ιρλανδική υπηκότητα. Οπότε Απευθύνω έκκληση, προσέξτε τη Ρεάλ Βιώνα. Δεν μπορείτε να την εμπιστεύετε. Ποτέ δεν κρατάει το λόγο της η Βρετανία, η Βρετάνια πάντα θα ε, αλλάζει τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρουτζίνσκι δεν βρίσκεται στην αίθουσα, οπότε πάμε στον Μικ Βόλας, επόμενο μιλητή. Δεν είναι ο προηγούμενος ομιλητής εδώ. Προφανώς ε, η αντιμετώπιση ε, των πολιτών στη, Ευρωπαίων στη Βρετανία και Βρετανών στην Ευρώπη πρέπει να ε, προστατευτεί. Ανεξαρτήτως του τι κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, τα δικαιώματα επίσης παρέχει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής πρέπει να διασφαλιστούν. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης την απειλή προς όλους τους πολίτες της νεοφιλελεύθερης ε, Ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε όρια στην εθνική διαδιοδότηση και οι διάφορες συμφωνίες ε, οδηγούν σε πολιτική λιτότητα που υπονομεύει τα δικαιώματα παιδείας, διατροφής, υγείας και στέγασης, καθώς και το δικαίωμα αξιοπρεπούς εργασίας, αμοιβή ε, και κοινωνικής ασφάλισης. Στην Ιρλανδία, ακόμη και αν είχαμε κυβέρνηση που θα είχε την οτροπία να αντιμετωπίσει την τρομακτική κρίση στέγασης που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, ε, θα του εμπόδιζαν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Με άλλα λόγια, η υποδομή μας, ε, οι οδοί μα, ε, χτίζονται από εταιρείε που την κάνουν να κοστίζει τρει φορέ παραπάνω χρήματα. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τροφοδοτεί και θρέφει τον ιδιωτικό τομέα με τι δικέ τη πολιτικέ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μου λείψει η Μαρτίνα από το Συνφέιν, αλλά θα μου λείψουν και οι συναδελφοί του κόμματος του Brexit. Θα λάμψουν τις αλλά πάντως εγώ είμαι υπέρ για το ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν ε, όσα προβλέπει η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Είδαμε τον Μπόρις του Τζόνσον να θριαμβολογεί και μας λέει ότι τώρα ξανά η συμφωνία γιατί εάν λειτουργεί η συμφωνία τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο στη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να συνεχίσουν να αποδεικνύουν ότι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αυτοκαθορισμού εάν θα φιωρούνται Ιρλανδοί, Βρετανοί ή τι οι Ιρλανδοί. Όλοι όσοι έχουν ε, ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να ε, βλέπουν να το δικαίωμά τους. Και τώρα για ένα λεπτό, κύριε Κιτσούκ, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων στην είναι στον Βασίλειο, γιατί πρόκειται για εκατομμύρια και είναι κάποιοι που έχουν υποβάλει αίτηση ε, διαμονής, προέρχονται και από τους 27 ε, κρατημέρια, γιατί υπάρχουν και οι Άγγλοι στην Ευρώπη, για να δούμε τι θα γίνει μετά την αποχώρηση. Οι πολίτες των 27 θα πρέπει επιγόντως να αποδείξουν ότι δικαιούνται να διαμείνουν στην χώρα μόλις λήξει μεταβατική περίοδος και η κυβέρνηση όμως της Αγγλίας θα πρέπει να σταματήσει να φέρνει προσκόμματα, να απειλεί με εκδίωξη από τη χώρα, γιατί αυτά φέρνουν αναταραχή. Ο Πρωθυπουργός Τζόνσον είπε ότι θέλει ε, στα τέλη του έτους να υπάρχει συμφωνία ομαλών σχέσεων. Όμως είναι θέμα ελεύθερης διακίνησης. Μετά το Brexit αυτό θα πρέπει να ισχύει, θα είναι σημαντικό και θα καθορίσει την μέλουσα σχέση. Λόπε Αγγιλάρ. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, τελικά καταφέραμε και ψηφίσαμε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μετά από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Με θλίψη βέβαια, γιατί θα μας λείψουν οι φίλοι μας οι Βρετανοί που είναι υπέρ της Ευρώπης. Δεν θα μας λείψουν όμως οι έδρες των λαϊκιστών, των αντιδραστικών που προκάλεσαν τον Brexit. Το μήνυμα όμως είναι σαφές. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριφερθεί στους Βρετανούς οι οποίοι κατοικούν στην Ευρώπη ανάλογα με τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στους Ευρωπαίους οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 30.000 ε, που είναι στα Κανάρια για παράδειγμα ή οι εργαζόμενοι που στην ε, Ισπανία 10.000 ε, κάθε μέρα πηγαίνουν στο Γιβραλτάρ και εργάζονται εκεί σε μια γωνιά της γης όπου υπάρχει ψωμένη η Βρετανική σημαία. Πολλή δουλειά όμως μένει ακόμα να γίνει για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα αυτά και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δέχεται την ε, ελεύθερη διακίνηση, τι θα γίνει με το άσυλο, την μετανάστευση, με τις αστυνομικές αρχές, πώς θα διασφαλίσουν την προστασία τόσο των Βρετανών στην Ευρώπη όσο και των Ευρωπαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστούμε. Χάναν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αυτή η συζήτηση φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα σε ένα παράλληλο κόσμο που δεν έχει και πολύ σχέση με την πραγματικότητα και με αυτά που συμβαίνουν. Εγώ πάντα ήμουνα επικριτικό στη στάση της Τερέσα Μέης και στην καθυστέρηση με την οποία αντιμετώπιζε το θέμα των δικαιωμάτων των ε, πολιτών, των Ευρωπαίων και των Βρετανών. Τώρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ των 27. Δεν είναι αλήθεια ότι αρνούμαστε. Δεν υπάρχει κανένα μηχανισμός να αρνηθούμε σε κανένα το καθεστώς του. Απλώς θέλουμε αποδείξεις. Αυτό μόνο. Και κάποιοι ήρθαν σε μένα επειδή φαινόντουσαν ε, σαν να μην μπορούν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους ε, κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι και ακούω του συναδέρφους να ζητούν ε, γραπτές μορφές ταυτότητας, όμως οι χώρες μέλη που δεν προσφέρουν την αμοιβαιότητα δεν επικρίνονται. Οπότε ποια είναι τα συμφέροντά τους, τι υποστηρίζουν τελικά. Ευχαριστούμε κύριε Χανέν. Μαρτίν Χόρουντ. Θέλω να πω ότι ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος ε, για τη Συμφωνία Αποχώρησης ε, επικρίνοντας το αυθαίρετο σύστημα του Ηνωμένου Βασίλειου που ήδη χειρίζεται άδικα ε, τους φίλους μας που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ήθελα να επανέσω τον Κίφερ Χόφστατ για τις τεράστιες προσπαθίες του να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών και των Βρετανών στα κράτη μέλη. Στην παράγραφο 20 το ψήφισμα αναγνωρίζει ότι πολλοί πολίτε ε, του ε, Βρετανοί που δεν θέλουν να χάσουν τα δικαιώματά του ε, ω Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να μπορέσουν να το διατηρήσουν. Εγώ το υποστηρίζω. Η ιδέα των διεθνών δικαιωμάτων για πολίτες ε, είναι κάτι υπαρκτό. Ε, θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει. Εμείς έχουμε δώσει δικαιώματα πολιτών ε, σε, σε πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας, όπως και στη Μάλτα, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της κοινοπολιτείας. Είναι κάτι λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε και θα παρεμποδίσει αυτή την τεράστια στέρηση δικαιωμάτων από σημερινούς Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστούμε για το όσα είπατε. Ο κύριος Αποσπισίλη είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του κειμένου και θεωρώ ότι ήταν σημαντικό το μήνυμα που στείλαμε. Μετά το Brexit, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων που κατοικούν στον Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να διασφαλιστούν. Είναι πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα και όταν κάποια στιγμή στο μέλλον δούμε τι λεπτομέρειε, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ισχύσει η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Να είναι θέμα προτεραιότητα. Είμαι Τσέχο. Είναι 35.000 οι μόνιμοι Τσέχοι, κάτι μόνιμοι κάτοικοι του Ιωμένου Βασιλείου. Άρα θα πρέπει να αποφασιστεί με ποιε προϋποθέσεις θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα του. πρόεδρου. Ένα λεπτό. Εγώ καταψήφισα το κείμενο για την αποχώρηση για δύο λόγους. Πρώτον, είναι φαρισαϊκό από το Βασιλείο να ξεκινά τέτοιες διαδικασίες υποδοχής όσων θέλουν να εγκατασταθούν στην χώρα λέει. Όμως είναι πολύ μπροστά, πολύ πιο μπροστά από τους 27 η χώρα όσον αφορά τα δικαιώματα. Χρειάζεται αμοιβιότητα γιατί υπάρχουν και οι Βρετανοί στην Ευρώπη δεν τα λέει αυτά το ψήφισμα. Δεύτερον, δεύτερος λόγος. Όταν το συζητήσαμε, αλλά και το κείμενο δεν λέει τίποτα για το δημοψήφισμα του 16. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με το Brexit. Πουθενά δεν αναφέρεται η σημασία του δημοψηφίσματος για τα όσα έγιναν. Πρόκειται για ακόμα μία ομή προσπάθεια ε, σαμποτάζ από πλευράς των Βρυξελών. Όμως το Κοινοβούλιο αποφάσισε και εγώ καταψήφισα. Νίνα η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα για να προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών μετά την αποχώρηση. Και πρέπει να είναι σαφέ το τι συμβαίνει στη μεταβατική περίοδο και τι συμβαίνει μετά τη μεταβατική περίοδο. Όπω ήδη ακούσαμε, υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια πολίτε Ευρωπαίοι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι έχουν ο καθένας τη δικιά του προσωπική ιστορία και προσωπική κατάσταση. Έχουν όμως και ένα κοινό ότι θέλουν να διασφαλίσουν τα, την προστασία τους, τα δικαιώματά τους για αυτούς και τις οικογένειές τους. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει τα πράγματα δύσκολα, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο όπως κάνει, που δεν προσφέρει ένα σύστημα που να τους εγγυάται απόλυτα να έχουν τα έγγραφα που τους χρειάζονται για να αποδείξουν ζητάνε έγγραφα από τους ιδιοκτήτες τους, από τους εργοδότες κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται έχω περιπτώσεις που αποδεικνύονται πολύ θλιβερές ιστορίες και εμπειρίες των Ευρωπαίων πολιτών που δεν καταφέρουν να τα έχουν όπως θα έπρεπε. Και παρόλο που προσφέρουν πολύ περισσότερα στο Ταμείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να ανησυχήσουμε και για το 1,2 εκατομμύρια Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τα δικαιώματα των δικών της πολιτών. Όσοι πάντως βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να ξέρουν ότι οι εργατικοί θα τους βοηθήσουν μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ακόμα χρόνο για άλλη μία εξήγηση ψήφου για το μέλλον της Ευρώπης θα συζητήσουμε δυστυχώς μόνο μετά από την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Οπότε στείλτε τα γραπτά ή παρουσιάστε τις εξηγήσει ψήφου αύριο μετά την ψήφο. Όπω είπα, λοιπόν, όποιε εξηγήσει ψήφου δεν μπορέσετε να παρουσιάσετε προφορικά, μπορείτε να τι υποβάλλετε γραπτό. Λοιπόν, μέλλον τη Ευρώπη, ε, λέω στου συναδέλφου που ενεγράφησαν για να μιλήσουν για αυτή τη συζήτηση. Δεν σα το λέω τώρα, δεν θα προλάβετε σήμερα το απόγευμα, γιατί μπορούμε να ασχοληθούμε με μόνο μία έκθεση ακόμα, αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την ετήσια έκθεση του 2018, Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο. Οπότε αυτοί οι συνάδελφοι να παραμένουν εδώ και επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Γιώνα Ομαρζέ για την ετήσια έκθεση του 2018 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την ευρωπαϊκή πολιτική επί του θέματος. Κύριε Ομαρζέ, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να απεικοδομήσουμε τους μηχανισμούς που παγκοσμίω οδηγούν σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αντιληφθούμε ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αποκλείεται να σταθούν όρθιες ε, παρά μόνο εάν χρησιμοποιούν απολυταρχικές πρακτικές και κάποια μορφή βίας που θεωρείται κυβέρνηση. Νεοφιλελευθερισμός και απολυταρχισμός είναι παράλληλα συστήματα. Αυτό αληθεύει στον κόσμο και στη Γαλλία επίσης, όπου παρατηρούμε πως ε, η σημερινή εξουσία ε, ε, μεταχειρίζεται με σκληρότητα τα κοινωνικά κινήματα. Βλέπουμε έκπληκτη και αδύναμη πως η εξουσία καταπνίγει τα κινήματα που θα έρθουν και θα αντιτεθούν στα φιλελεύθερα προγραμματά του. Σήμερα στη Γαλλία ο θάνατος περιμένει ε, ειρηνικούς διαδηλωτές. Η αστυνομική βία πολλαπλασιάζεται και χρησιμοποιείται για την τήρηση της τάξης με χρησιμοποιώντας όπλα ε, που έπρεπε να χρησιμοποιούνται κανονικά σε πόλεμο και που απαγορεύονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Σήμερα στη Γαλλία ε, διαδηλωτές, δημοσιογράφοι συνδικαλιστές υποχωρούν και μαζί με αυτούς υποχωρούν και οι ατομικές ελευθερίες που ωστόσο ε, θεσπίζονταν και στο δικό μας σύνταγμα και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αναρωτιέται κανείς καθώς ε, οι αρχές διαδοχικά πλήττονται, ε, απορρίπτουμε αξίες, ασκούμε υπερβολική εξουσία. Τι Γαλλία διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή σιγά σιγά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, τηρείτε το χρόνο για να μπορέσουμε να προλάβουμε να τελειώσουμε στην ώρα μας. Η κυρία Σόιντροβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πάντα να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αποτελεί συνήγορό τους παντού στον κόσμο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να θυσιάζονται ε, στο όνομα των επιχειρήσεων και των business. Πρέπει να υπάρχουν σωστά κίνητρα στην αναπτυξιακή βοήθεια και να στηρίζουμε τις κυβερνήσεις εκείνες που προσπαθούν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες τους. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στην κατάσταση των χριστιανών. Δυστυχώς δεν εγκρίθηκαν αυτές οι τροπολογίες. Πρόκειται για χριστιανούς οι οποίοι συχνά αποτελούν στόχο διακρίσεων και βίας. Και δεν γίνεται καμία έκκληση ε, τελικά για να προστατευτούν. Αναρωτιέμαι πόσο σοβαρό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά επ' αυτού. Γι' αυτό και στο τέλος καταψήφισα το ψήφισμα. Ευχαριστούμε. Ε, ούτε ο κύριο Πόλτσακ είναι εδώ. Ε, η κυρία Ντέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά κανονικά ε, και αδιέρετα. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί κανείς. Αλλά δυστυχώς αυτό κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανακατεύουμε με την πολιτική μας και τα βάζουμε τις χώρες που δεν μας αρέσουν ή κυρίως εκείνες που δεν αρέσουν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Με παράνομους τρόπους, με εδώ, εδώ πέρα με την δολοφονία του Σελεϊμάνη και τον Αμπούλ Μαρτζή Μοχαντές του Ιράκ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει, σιωπά απέναντι σε αυτά θα έπρεπε να είχαμε το θάρρο να τολμήσουμε να μιλήσουμε παντού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ πέρα πρόκειται για ε, στρατηγού οι οποίοι εκτελούνται σε μια κυρίαρχο χώρα που είναι το Ιράκ. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα λέγαμε αν οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο δικό του επικεφαλή του προσωπικού, για παράδειγμα, είχε δολοφονηθεί από του Ρώσου. Πολλά θα λέγαμε τότε. Αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα με αυτή την έκθεση. Μιλάμε, μιλάμε, μιλάμε, καταδικάζουμε αυτού που δεν μα αρέσουν και δεν λέμε τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι παραβιάσει του αλλού. Η βία της γαλλικής ε, σημερινή κυβέρνηση απέναντι σε ειρηνικού διαδηλωτέ, Τι σα λέει, τα είπε και ο συνάδελφο ή με τους Καταλανού που δεν του αφήνουμε να πάρουν την έδρα του εδώ. Γι' αυτό και εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστούμε για την άποψή σας. Τώρα στα νογκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ούτε εγώ είμαι υπέρ της επιμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κουνάει το δάχτυλο στο τι θα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαιούμεθα να επιπλήσουμε τους άλλους όταν οι ίδιοι είμαστε άριστοι μαθητές, πρωταθλητές στο μέλλον των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά, εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματο. Μόνο και μόνο γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική παράγραφος εκεί που αναφέρει το πρόβλημα των απατριτήτων, οι οποίοι απάτρε θα πρέπει μέχρι το 24 να έχουν βρει κάποια λύση εντός και εκτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και για την χώρα με την ε, Λετωνία. Ε, γιατί οι απάτριδες στη χώρα μας δεν μπορούν να ψηφίσουν, δεν έχουν πολλά άλλα δικαιώματα. Βέβαια, το ίδιο και για αυτούς που με άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και λόγω της προέλευσής τους έχουν χαρακτηριστεί απάτριδες. Οι περισσότεροι είναι ντόπιοι. Όμως αυτό είναι δυσμενής διάκριση επί τη βάση της ε, προέλευσης. Αυτό το λέει το κείμενο, κρίμα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γέρζη τελευταίος για αυτή την έκθεση. Και κατόπιν έχουμε ακόμα δύο μικρές εκθέσεις και μετά το κείμενο για το μέλλον της Ευρώπης. Θα το πούμε αύριο. Κύριος Πόσπισιλ, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου, διότι θεωρώ ότι η υπόθεση των το δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντική για την ε, Ένωση και θα πρέπει βέβαια να προσέχουμε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, έχω μια παρατήρηση, παρά το ότι υπερψήφισα. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να μείνουν ωραία λόγια. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η Επιτροπή όλα αυτά να τα υλοποιήσει. Υπάρχουν κάποιε χώρε στις οποίες ε, παρέχεται οικονομική βοήθεια. Ε, θα πρέπει αυτή η βοήθεια να εξαρτηθεί από την τήρηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Να μην υποστηρίζουμε ε, χώρες που έχουν κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μείνουν όλα αυτά ωραία λόγια. Θα δούμε τώρα την έκθεση του David McAllister για την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Έχουμε τρεις ομιλητές. Την κυρία Σόιντροβα, εκ μέρους του ΕΛΚ, η πρώτη ομιλήτρια. Έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει την ε, ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας ε, σε πολυμερή βάση σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί τη βασική εγγύηση για την ασφαλεία μας, σίγουρα. Και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Εγώ είχα κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το κομμάτι που αφορούσε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. που υποτίθεται ότι θα ήταν ο τρίτος πυλώνας της πολιτικής αυτής. Ε, πιστεύω ότι στο τομέα αυτό θα πρέπει να έχουμε κυρίαρχο ρόλο του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση αυτή για την ε, πολιτική αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βρετσιόνοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω τη στάση μου προς αυτή την εκθέση την οποία δεν υποστήριξα. Αφενός περιγράφει πολύ όμορφα η έκθεση της προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε όσον αφορά την ανάγκη μιας πιο αποφασιστικής αντιμετώπισης της Ρωσίας, όσον των απειλών στον κυβερνοχώρο και των λοιπόν απειλών με τις αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω για την ε, ε, διέλευση από τα σύνορα και καλών και κακών ανθρώπων. Κάποιοι απλά θέλουν να έρθουν για να ε, ζήσουν ευημερία, για να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή και άλλοι θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές της, να ε, διαπιστώσει επιτέλους ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι απειλή και το Ισραήλ είναι ένα σύμμαχος. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν αλλαγή. Αυτό μου έλειψε από την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, καταψήφισα την έκθεση διότι είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατά της εισόδου Ρουμανίας και Βουλγαρίας, ε, κατά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Έχει τρομακτικές ε, αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία τρομακτικές συνέπειες για τη δική μου χώρα, για τη Γερμανία. Οδήγησε σε πορνεία, οδήγησε σε έγκλημα, υπο... νόμευσε την κοινωνική διάσταση στην περιοχή του Ρούρ στη Γερμανία. Είναι φρικτές οι συνέπειες για μας και το βλέπω όχι μόνο εγώ, το λένε το λέει και ο δήμαρχος ε, του Ντόρτμουντ ε, και άλλων πόλεων που είναι σοσιαλιστές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι λιγότερη ελεύθερη κυκλοφορία, όχι περισσότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ωραία. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση μέχρι τις 3 διακόπτουμε. Στις 3 το απόγευμα θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. puhemies Hyvää iltapäivää. Istunto jatkuu. Η πρόεδρος. Ξαναρχίζει η σύνοδος, λέει η πρόεδρος. Αλλά πρώτα πρώτα να εγκρίνουμε τα χθεσινά μας πρακτικά. Υπάρχει κάποια ένσταση, κάποια παρατήρηση επί των πρακτικών. Όχι από ό,τι φαίνεται, οπότε θεωρώ ότι εγκρίνονται. Και πάμε εδώ στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο ουσιαστικό θέμα είναι ε, συζήτηση επίκαιρου θέματος διαστρέβλωση της ευρωπαϊκής ιστορίας και μνήμη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι στην λόγο συζήτηση δεν πρόκειται να δοθούν ε, επιπλέον ε, θέσεις ε, και χρόνους αγορεύσεως ή μπλε κάρτες. Κύριε Βέμπερ, έχετε το λόγο. Κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται περί της ιστορίας. Συζητούμε τώρα το μέλλον μας, διότι εάν κανείς αγνοεί την ιστορία του, τότε παραμελεί το μέλλον του. Μιλούμε για περισσότερα από 40 εκατομμύρια νεκρών. Αυτοί μας λένε ποτέ πια. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο έγκλημα. Ξεκίνησε η ναζιστική Γερμανία αυτόν τον πόλεμο και αυτό έφερε ως τίμημα αποτρόπια εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητος. Κάθε Γερμανός πολιτικός θα πρέπει να αναλάβει για λογαριασμό της χώρας μας τις ευθύνες του. Όμως κάθε πολιτικός εντός και εκτός της Ευρώπης επίσης φέρει την εξή ευθύνη. Να μην παίζει, μην χειραγωγεί την ε, ιστορία. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν δέχεται την προσπάθεια αναθεώρησης ιστορίας από τον Πούτιν. Θα πρέπει βεβαίω να ξεκαθαρίσουμε ότι επιτέθηκε η Ναζική Γερμανία στη Ρωσία και υπέφερε ε, κατά τον πόλεμο. Αλλά θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι υπήρχε το σύμφωνο Χίτλερ και Στάλιν. Δύο δαίμονες, δύο αποτρόπαιοι δικτάτορες. Αυτή η συμφωνία Χίτλερ-Στάλιν ήταν η αρχή του κακού για πολλές χώρες. Πολωνία, Φινλανδία, Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία και Ρουμανία που υπέστησαν την επίθεση. Αυτό το σύμφωνο σήμαινε ότι εκατομμύρια Ευρωπαίων σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ε, χτυπήθηκαν επί δεκαετίες με καταπίεση δικτατορία. Επρόκειτο για ένα σύμφωνο έγκλημα κατά ειρήνης και δημοκρατίας. Έχουν περάσει από τότε 80 χρόνια και παραπάνω. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ποτέ πια σήμερα στην Ένωση και στο ΝΑΤΟ τιμούμε την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ελευθερία και για την κεντρική και ευρωπαϊκή Ευρώπη, όλοι ενωμένοι, αλληλέγγυοι στην Ευρώπη, με την μνήμη την ιστορική, για να προστατεύσουμε το μέλλον, που είναι κοινό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέμπερ. Τώρα θα ακούσουμε το Συμβούλιο. Νικόλινα Γιάσκη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή που μου δίνετε να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Πράγματι, άκουσα και αναγνωρίζω τι ανησυχίε που εξέφρασε ο κύριο Βέμπερ και γνωρίζω πολύ καλά σε τι αναφέρεται που έχει να κάνει με τις πολωνικές αρχές. Θέλω εδώ να εκφράσω την ε, συμπαθιά μου προς όλα τα θύματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Πράγματι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει η Ευρώπη αν θέλει να αντιμετωπίσει το μέλλον της. Η σημερινή συζήτηση μας προβληματίζει για το πώς μαθαίνει η Ευρώπη από την ιστορία τη